μετά την ε, παρουσίασή σας και κλείνει η συζήτηση τη Τετάρτη στις 12 θα γίνει η σχετική ψηφοφορία. Θα ήθελα να σας ε, πω κυρίες και κύριοι ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο στις 11 Μαρτίου 2013, 8.30 το πρωί έως τις 2 και μετά μεταξύ 3 και 11 το βράδυ. Έχετε στο ε, στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου την ατζέντα και έτσι λοιπόν διακόπτεται η σύνοδος. Καλή νύχτα